Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε. Τη διάσκεψη των Προέδρων, την ανοιχτή διάσκεψη των Προέδρων. Otwieram posiedzenie Λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση της διασκέψεως των Προέδρων. Θυμίζω ότι είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου η συνεδρίαση αυτή. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους, να καλωσορίσω τον κύριο Βανρόμπα και τον κύριο Μπαρόσου τον πρόεδρο λοιπόν του Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, πήραν μέρος στις τελευταίες συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έμεινε στην ιστορία σαν ένα από τα κομβικά θα έλεγα σημεία της ιστορίας του Συμβουλίου. Ξέρουμε τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν Ξέρουμε ότι υπήρχαν ε, ε, δύο ακαθόδη θέματα. Πρώτον το θέμα του Σέγγεν και δεύτερον η κρίση του ευρώ. Το ευρώ σαν νόμισμα και το Σέγγεν σαν χώρος ελεύθερης διακίνησης είναι δύο θα έλεγα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να προστατευθούν προσεκτικά. Έχουμε ξεκάθαρη άποψη για αυτά τα δύο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό η συνάντησή μας εδώ σήμερα είναι σημαντική. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Βαν Ρόμπαϊ και τον κύριο Μπαρόσο που βρήκαν τον χρόνο στη δύσκολη αυτή περίοδο να είναι μαζί μας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Βαν Ρόμπαϊ θα μας μιλήσει για τα συμπεράσματα της προηγούμενης εβδομάδας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τιμή είναι να σας αναφέρω αυτά τα οποία αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου σημειώθηκε πρόοδο σε αρκετά θέματα. Την πρώτη μέρα την αφιερώσαμε στην οικονομία, στα οικονομικά θέματα είχαμε τις εξής αποφάσεις. Συντονισμό της οικονομικής πολιτικής πρώτα με το, έτος, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες. Δεύτερον το πλήρες πακέτο και τρίτον η κατάσταση χωρών και όσον αφορά το πρόγραμμα για το IMF συμπεριλαμβανομένων αυτών των χωρών. Πρώτο τμήμα, πολιτική συντονισμού, οικονομική πολιτική συντονισμού. Ολοκληρώσαμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό. Είχαμε καλή και μακρά συζήτηση για τις εθνικές δημοσιονομικές επιλογές και τους τρόπους και υιοθετήσαμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα κράτη-μέλη χωρίς, το τονίζω, χωρίς να αποδυναμώσουμε αυτές τις προτάσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τόσο περισσότερο μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πραγματικά στεναρές συστάσεις ε, και προτάσεις. Και τώρα είναι δουλειά των κρατών μελών. Αυτές οι συστάσεις πρέπει να τις λάβουν υπόψη όταν θα συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους και όταν θα καταρτίζουν προγράμματα μεταρρύθμισης και αναθεώρησης. Αυτό το οποίο έχω συναγάγει από τις συζητήσεις μας είναι όχι μόνο ότι μπορούν να γίνουν δεκτές από τα κράτη-μέλη συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει και να εφαρμοστούν. Επίσης ζητήσαμε και τις δεσμεύσεις ε, υπό το σύμφωνο Europlus σε σχέση με όσους συμμετέχουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όλοι συμφωνήσαμε από αυτόν και εργαζόμαστε στη σωστή κατεύθυνση τονώνοντας τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα, τις ε, ε, μεταρρυθμίσεις και τον τομέα συνταξιοδότησης συντάξεων ώστε να είμαστε βιώσιμοι στην οικονομική μας προσπάθεια. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξο το πλαίσιο δράσεων στο μέλλον. Με αυτή τη στεναρή ε, πολιτική μαθημάτων έχει συναγάγει τα συμπεράσματά της η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ε, δημοσιονομικά θέματα. Οι αποφάσεις σε μια χώρα έχουν επιπτώσει σε όλες τις άλλες, ε, ιδιαίτερα σε εκείνες ε, που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα, στο ευρώ. Αυτή η πρώτη εμπειρία είναι θετική. Υπάρχει εντονότερο αίσθημα κοινή ευθύνη. Ακόμα και αν αυτές είναι κρίσιμες ημέρε σε περίοδο κρίσης τονώνουμε το πλαίσιο το δημοσιονομικό. Δεύτερο στοιχείο στα οικονομικά θέματα που συζητήθηκαν. Το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά το περιεκτικό πακέτο των οικονομικών μέτρων. Εδώ υιοθετούμε το αναθεωρημένο κείμενο για την ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Μέσο Σταθερότητας και τον μηχανισμό Ευρωπαϊκής Νομισματικής Σταθερότητας για το μέλλον. Έχουμε και αναγνωρίζουμε τον ρόλο κλειδιού που έχουν οι τράπεζες και το τονίζουμε αυτό. Βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο τονώνοντας την οικονομική διακυβέρνηση. Ένα ισχυρότερο σύμφωνο σταθερότητας και μια νέα μακροοικονομική εποπτεία. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για αυτά τα σημεία που γνωρίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το έργο που επιτελείτε εσείς. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν σε παραπάνω από 95% των διατυπώσεων του κειμένου και γι' αυτό απευθύνω έκκληση στους νομοθέτες να ολοκληρώσουν τις τελικές διαπραγματεύσεις ώστε αυτό το σημαντικό πακέτο να μπορεί σύντομα να εγκριθεί και ελπίζω πράγματι στην επόμενη κοινοβουλευτική συνεδρίασή σας. Συγχαίρω την Ουγγρική Προεδρία και το Κοινοβούλιο για το έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε σημαντικές βελτιώσεις. Σύμφωνα με τον Ούγγρο Υπουργό Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, η ποιότητα του κειμένου βελτιώθηκε σημαντικά. Το πακέτο έγινε πιο ισχυρό και πιο συνεκτικό. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο κατάφερε μεταξύ άλλων τα εξής να τυποποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα νομοθετικά κείμενα και πρόβλεψη για την αξιολόγηση των κρατών μελών, ευρεία αξιολόγηση για την στρατηγική του 2020 για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, να διασφαλιστεί ότι αντίστροφη ειδική πλειοψηφία θα εφαρμόζεται σε πέντε από τις έξι αποφάσεις όπου αυτό θα είναι νομικά εφικτό, ακόμα και των συστάσεων όσον αφορά την επανόρθωση και την ε, διόρθωση των ε, ανισορροπιών ε, στις μακροοικονομικές συνιστώσεις. Και εδώ υπάρχει και η δυνατότητα που προσφέρει το Συμβούλιο για τη ρήτρα διάσωσης. Επίσης, να διαδραματίζει ισότιμο ρόλο το Κοινοβούλιο εναντί του Συμβουλίου για τον πύχη των επιδόσεων, τον κατάλογο επιδόσεων στις μακροοικονομικές αυτές αξιολογήσεις. Τη της, ε, ε, της διαφθοράς, εισαγωγή νωρίς κυρώσεων όταν θα υπάρχουν υπερβολικές υπερβάσεις Αυτά δεν είναι συνηθισμένα πράγματα και ίσονο σημασία, αλλά σημαντικά. Και προ το ε, Κοινοβούλιο αλλά και προ το Συμβουλίο θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να επιτευχθεί συμφωνία σε ένα καλό συμβιβασμό. Οι θέσει βρίσκονται πολύ κοντά η μία προ την άλλη και γνωρίζω ότι περαιτέρω οποιασδήποτε άλλε σημαντικέ αλλαγέ θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όπως ε, λένε στα γαλλικά, δεν θα πρέπει το καλύτερο να είναι ο εχθρός του καλού. Και το επαναλαμβάνει στα αγγλικά ο κύριος Φαν Το τρίτο και το τμήμα που ολοκληρώνει αυτό το πακέτο για τα οικονομικά θέματα είναι η κατάσταση των χωρών υπό το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καλωσορίζει την πρόοδο στην Ιρλανδία το Συμβούλιο για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται σε καλή πορεία. Επίσης, καλωσόρισε την διακομματική συμφωνία στην Πορτογαλία πλήρως να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και όσον αφορά την Ελλάδα, υιοθετήσαμε ένα περιεκτικό ευρύτερο κείμενο, το οποίο θα έχετε δει στα συμπεράσματα. Υπογραμμίζεται η απόλυτη σημασία που δίνουμε στην έγκριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Ελλήνων, των κύριων στρατηγικών της δημοσιονομικής πολιτικής. Η Βουλή των Ελλήνων εξετάζει σήμερα ακριβώς αυτά τα θέματα. Η έγκριση τους θα δημιουργήσει τη βάση για την κοινή υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους και το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα δώσει τη δυνατότητα έγκαιρα να καλυφθούν τον Ιούλιο οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ελλάδας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ευρώ υιοθέτησαν τις αποφάσεις ε, όσον αφορά την 20η Ιουνίου για την παρακολούθηση, την συμμετοχή ε, του ε, ιδιωτικού τομέα εθελοντικά όσον αφορά στο χρέος ε, ε, ακολουθώντας ε, την οδό της δημοσιονομικής ανακούφισης. Επικεντρώσαμε τη συζήτησή μας σε τρία θέματα. Απάντησή μας στις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο, μετανάστευση και ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας. Για το πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να συνεχίσει να διαδραματίζει ιστορικό ρόλο στις ιστορικής σημασίας εξελίξεις που τεκταίνονται στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή χωρίς την Ευρώπη θα υπήρχε μια ευρωπαϊκή, μια αραβική, ε, με συγχωρείτε, άνοιξη, αλλά χωρίς αμφιβολία δεν θα οδηγούσε σε ένα ε, αραβικό θέρος. Και σε σχέση με τις ε, δημοκρατικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στην Αίγυπτο και στην Τινησία βλέπουμε και τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στο Μαρόκο, νέες προσπάθειες στην Ιορτανία και την άρση της κατάστασης πολιορκίας στην Αλγερία. Θέλουμε να συνεισφέρουμε υπέρ όλων αυτών των αλλαγών και προσφέρουμε μια νέα εταιρική σχέση στις χώρες της περιοχής αυτής, προωθώντας και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών τους αξιολογούμε τις ε, επιδόσεις ε, των εταίρων και τις ανάγκες τους. Ε, <clears throat> λιγότερα για λιγότερα, περισσότερα για περισσότερα. Και ως Συμβούλιο <clears throat> καταδικάζουμε την καταστολή και την ομή βία Συρία και συνεχίζει το καθεστώς στη Συρία δυστυχώς να ασκεί αυτή την ομίβια εις βάρος των ίδιων των πολιτών της. <clears throat> αντί να υλοποιεί τις υποσχέσεις της για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις ακολουθώντας μια πολιτική καταστολής αμφισβητεί την ίδια τη βάση στην εξουσία της η κυβέρνηση της Συρίας, το καθεστώς Συρίας. Τέτοιου είδους περιπτώσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στο να προσταθούν στη δικαιοσύνη υπεύθυνοι και σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την 20 Ιουνίου 2011 καλωσορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υιοθέτηση και έγκριση νέων κυρώσεων και δίνει πλήρη υποστήριξη στις διπλωματικές προσπάθειες που θα διασφαλίζουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνες, ευθύνες του και να δώσει επαρκείς απαντήσεις στην κατάσταση στην Συρία. Όσον αφορά την Λιβύη θα συνεχίσει να υπάρχει η στρατιωτική πίεση εις βάρος του καθεστώτος τη της Λιβύης εφόσον συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία. Όσον αφορά την Ιεμένη, επαναλαμβάνουμε ότι είναι κατεπήγον να μπορέσει να διασφαλιστεί η μεταβατική δημοκρατική περίοδος. Το δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε κάτι δεύτερη ημέρα είναι η μετανάστευση επελέγει αυτό το θέμα και προηγούμενα πριν από την Αραβική Άνοιξη και είναι κατεπήγον να υπάρξουν συμπεράσματα. Πρώτο συμφέρον, να ανακουφιστεί η πίεση στα νότια σύνορά μας, βοηθώντας τους νέους στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή να υπάρξει ένα θετικό μέλλον για αυτούς στις χώρες τους. Μια επιτυχής πολιτική μετανάστευση ξεκινά έξω από τα σύνορά μας. Γι' αυτό οι νέες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη της νότιας γειτονίας, γειτονιακής σχέση, θα συμπεριλαμβάνουν τα θέματα μετανάστευση και ασφάλεια. Δεύτερον, σε αυτό το άσυλο, είπαμε ότι σε σχέση με τι διαπραγματεύσει του Συμβουλίου θα πρέπει να, να επανεξεταστούν οι νέε προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσει. Και επιβεβαιώνουμε ότι ο ε, στόχος του 2012 ισχύει για την θέσπιση μιας κοινή ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επιπλέον για το Σέγγεν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύονται απόλυτα για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Είναι θεμελιώδους σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα θεμελιώδες δικαιώμα των πολιτών. Χωρίς να υπονομευθούν αυτές οι αρχές υπάρχει ανάγκη να τονωθούν οι κανόνες του Σέγγεν. Ρήτρες ασφάλι, διασφάλισης θα πρέπει να εισαχθούν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ανταποκριθούμε σε ειδικά γεγονότα όσον αφορά την ε, υπονόμευση της, ε, των αρχών της Συμφωνίας ε, Σέγγεν χωρίς να διακυβεύεται όμως η ελευθερία κυκλοφορίας πολιτών. Ως τελευταίο μέτρο, ίστατο μέτρο, μέσα στο πλαίσιο αυτών των ρητρών μια ρήτρα θα μπορούσε να εισαχθεί που θα επιτρέπει την έκτακτη εισαγωγή συνοριακών ελέγχων για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης κατάστασης όταν δεν είναι βέβαιο ότι ένα κράτος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Με συγκεκριμένα στοχοθετημένα κριτήρια θα λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση και με μια κοινή αξιολόγηση αυτών των στόχων και της περίοδου κατά την οποία θα ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε έγκαιρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Υιοθετούμε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ενίσχυση της Frontex, της υπηρεσίας μας ε, για τα εξωτερικά σύνορα. Θα επιτρέψει αυτό την Frontex να αναπτύξει συνδέσμους αξιωματούχους ε, από κοινού με την πολιτική γυτνίασης με τα γειτονικά μας ε, κράτη. Και τώρα η Ευρωπαίοι συνοριοφύλακες σε ομάδες θα συνεχίσουν αυτό το έργο. Και τέλος συζητήσαμε το θέμα της Κροατίας. Προλιάνθηκε το έδαφος για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένουμε το Συμβούλιο να ολοκληρώσει πολύ σύντομα τις διαπραγματεύσεις που εκκρεμούν πριν από τα τέλη Ιουνίου. Μετά θα υπογράψουμε τη Συμφωνία Ένταξης και όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ένταξη θα γίνει κατά τα μέσα του 2013. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια νέα προώθηση στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Πέρα από όλες αυτές τις συζητήσεις πολιτικών θεμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε τον κύριο Μάριο Ντράγκη ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την 1η Ιουλίου εφέτος. Μετά από την ευνοϊκή γνώμη που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά ολοκληρώνουν την εισήγησή μου και έκθεση επί διαφορετικών θεμάτων για ένα εργασία, ε, τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για την απόφαση για την Κροατία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση απομένει η υλοποίηση μιας μεγάλης φιλοδοξίας που τώρα θα ευδοκιμήσει. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ζητήσω τώρα από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε ένα πολύ ουσιαστικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πήρε αποφάσεις που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέραμε εδώ στην οικονομική πολιτική, τη μετανάστευση, την Νότια Μεσόγειο και την ένταξη της Κροατίας για την κατάσταση στην Ελλάδα για μια ακόμη φορά δείξαμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε όταν απαιτείται να υπάρξει συμφωνία και χαίρομαι να αναφέρω ότι η εφαρμογή του προγράμματος μαζί με το Δέλτα Νιτάφ στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία πηγαίνει καλά. Εμείς σε καθημερινή βάση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αλληλοσύνδεσής μας θα έλεγα αρκετούς μήνες μετά από την υιοθέτηση του πακέτου, ο στόχος της παρέμβασης έχει πλέον τεκμηριωθεί. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σωστά τον τρόπο αντιμετώπισης της αλληλοεξάρτησης των οικονομιών μας με μια πραγματική οικονομική πολιτική στην Ευρώπη και στην περιοχή του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την αποκατάσταση των δημοσιονομικών και υπάρχει δυνατότητα όπως διευκρίνησα μιλώντας για την Ελλάδα, να παίρνουμε εκ των προτέρων μέτρα τα οποία να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφασή μας να προκαταβάλουμε ουσιαστικά χρήματα και να δώσουμε και τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα για να συνοδεύσουμε έτσι κάποια μέτρα αναπόφευκτα, μερικές φορές οδυνηρά, τα οποία προσφέρουν και αυτά με τη σειρά τους προς την ανάπτυξη. Νομίζω ότι η συνεισφορά της Επιτροπής και οι προτάσεις της προσυζήτηση ήταν πολύτιμες στις συζητήσεις του Συμβουλίου και ήταν θα έλεγα η βάση για τους ξεκάθαρους προσανατολισμούς που θα μας κατευθύνουν τους επόμενους μήνες. Προχωρούμε προς μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για την Ευρώπη Υπολογίζω λοιπόν στη συνεργασία των συνομοθετών έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε πλήρως το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητά μέλη, εντυπωσιάστηκα από την ειλικρίνεια των συζητήσεων ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στις συστάσεις των διαφόρων κρατών που οδήγησαν στις συνενέσεις και τους συμβιβασμούς. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονταν μέχρι τώρα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αναγνωρίζουμε με πρακτικούς όρους την αλληλοεξάρτηση των οικονομιών μας και να αποδεχθούμε να κάνουμε μια ποιοτική προσπάθεια στον τομέα της λήψης αποφάσεων. Οι συζητήσεις αυτές χαρακτηρίζονται όλες από μια επίδειξη καλής βούλησης θα έλεγα η οποία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο προς τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει και στον τομέα της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Υπάρχει ανάγκη μείωσης του βάρους του γραφειοκρατικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει και ένα οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς το 2015. Η πρόοδος προς τους στόχους της στρατηγικής του 2020 είναι σημαντική, αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε επί τη βάση των ανακαινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί γιατί υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει σωστά. Φυσικά δεν έχουμε ψευδεστήσεις σε σχέση με τις δυνατότητες προόδου, όλα εξαρτώνται από την εθνική εφαρμογή των μέτρων αυτών. και από την ένταξη του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου στα εθνικά εξάμεινα τα οποία έχουν γίνει πλήρως δεκτά φυσικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η μετανάστευση, και αυτό δεν εκπλήσει επίσης κανένα, δημιουργεί πάρα, πολλά, πάρα πολύ, ε, θα έλεγα, πάρα πολύ ενδιαφέρον στις συζητήσεις. Μερικές φορές τα θέματα της μετανάστευσης χρησιμοποιούνται και από εξτρεμιστές λαϊκιστικές δυνάμεις κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κατά της παράδοσης των δημοκρατικών κοινωνιών της Ευρώπης. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να διαχειριστούμε τα θέματα της μετανάστευσης. Είπα πολλές φορές και θα το ξαναπώ ότι η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων είναι ένα βασικό θα έλεγα έκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πυλώνας της δραστηριότητάς μας και είναι κάτι το κρίσιμο στα πλαίσια της οικονομικής ανάκαμψης. Δεν θέλουμε λοιπόν την ελευθερία διακίνησης και τις βασικές αρχές της ελευθερίας κυκλοφορίας και διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τίθενται σε αμφισβήτηση. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν η πλήρης αναγνώριση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη ελεύθερη διακίνηση των προσώπων σαν κεντρικό χαρακτηριστικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θεμελιώδε δικαίωμα των πολιτών τη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια τη συζήτηση για τη μετανάστευση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να προστατεύσουμε το Σέγγεν, πρέπει να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση του Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει νέες προτάσεις για μια σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης. Αυτό έγινε δεκτό λοιπόν και από το Συμβούλιο και είναι μια αρχή που εδράζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμπληρώσουμε το σύστημα αυτό με ένα σύστημα εγγυήσεων που δίνει τη δυνατότητα κάποιων επιπλέον ανταποκρίσεων στις ε, απειλές και στις καταστάσεις όταν τα εξωτερικά μας σύνορα υφίστανται σοβαρές πιέσεις. Σαν ίστατη θα έλεγα παρέμβαση μπορούν τα κράτη-μέλη να αποκαταστήσουν τους εξωτερικούς τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός αυτός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα εφαρμογή την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών μεταξύ των οποίων την ελεύθερη διακίνησή τους. Για το άσυλο είναι ξεκάθαρη θέση μας. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το κοινό μας σύστημα μέχρι το τέλος του 2012. Για να το πετύχουμε αυτό κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι υπάρχει η όθηση για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Η πολιτική μας για την γειτονία προς τον Νότο συζητήθηκε. Επίσης το Συμβούλιο υποστήριξε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ της Εκπροσώπου για την υποστήριξη της δημοκρατίας και της ευημερίας των χωρών του Νότου της Μεσογείου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου παρουσίασε τα αποτελέσματα αυτά, οπότε δεν θα μείνω στις λεπτομέρειες. Θα στραφώ τώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου υπήρξε μια ιστορική απόφαση για την ένταξη της Κροατίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο τέλος του μήνα, έτσι ώστε να υπογραφεί η ένταξη μέχρι το τέλος του 2011. Η διαδικασία η ενταξιακή χαρακτηρίστηκε από ε, αυστηρές προϋποθέσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κροατία να διατηρήσει τις μεταρρυθμιστικές της προτάσεις για να προετοιμαστεί για ένταξη. Και θα ήθελα να βοηθήσουμε έτσι στην αποκατάσταση της ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια. Μια τελευταία λέξη για την Ελλάδα. Έχουμε ένα σχέδιο για την Ελλάδα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγική που εγκρίθηκε από τη λεγόμενη Τρόικα σε συνεργασία με τι ελληνικέ αρχέ. Χρειάζεται τώρα η Ελληνική Βουλή να διπλασιάσει τι προσπάθειές τη για να επιβάλλει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσεις. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι και αδιέξοδη. Χρειάζεται αποφασιστικότητα για να πράξουμε πάνω δυνατό για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βαδίσει πάνω σε αυτή την δύσκολη ατραπό όπου βρίσκεται για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της που είναι και το κλειδί για την μακροπρόθεσμη ευημερία της χώρας αυτής. Στις δύσκολες στιγμές προσπάθειας αυτής θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε μια κοινωνική ευθύνη. Δεν θα πρέπει να φοβηθούμε τις δύσκολες αλλαγές, αλλά να μην λησμονούμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε για την επιστροφή του χρέους για τα τοκοχρεωλήσια και τους τόκους είναι ένα ευρώ που δεν μπορεί να πάει για νοσοκομεία, για δρόμους, για δημιουργία απασχόληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις ε, βαθιές ε, δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να προχωρήσει στον δρόμο της ανάπτυξης. Τέλο, συγχαρητήρια στον Μάριο Ντράγκη για τον διορισμό του ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τραπέζη από τον Νοέμβριο Φέτο, Πρόκειται για άνθρωπο αφοσιωμένο στα ευρωπαϊκά ιδιώτη και ε, απόλυτα καταρτισμένο σε όλα τα σχετικά με την οικονομία θέματα. Του ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία στο έργο του και πιστεύω ότι έχουμε πλέον με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια βάση για να προχωρήσουμε στα πολύ κρίσιμα θέματα της ε, οικονομικής διακυβέρνησης καθώς και της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος Μπούσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις παρατηρήσεις σας, για την ε, ομιλία που εκφωνήσατε εξ ονόματος τώρα των ε, πολιτικών ομάδων για το Λαϊκό Κόμμα πρώτα. Ο πρόεδρος κύριος Ζωζεφ Ντόλ. Έχετε το λόγο κύριε. Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και οι άλλες χώρες, οι υπερχρεωμένες χώρες που τιμωρήθηκαν από τις αγορές τελευταία, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Χαίρομαι που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνειδητοποίησαν το γεγονό αυτό και κατέληξαν σε ενιαία θέση στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την οικονομία, για τη μεταναστευτική πολιτική, καθώ και για τι σχέσει μα με του γείτονε προ Ανατολά και προ Νότον. Το επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει εξ ονόματο τη ομάδα μου, ότι από την αρχή τη κρίση είπαμε ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Μα σα παρακαλώ, κύριε Φαράντ, Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα σα επιτρέπει να αποχωρήσετε, εσείς και η χώρα σας. Κανένα δεν πρόκειται να θρυνήσει. Είναι σαφέστατο αυτό. Έτσι είναι. Για το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, χρειάζονται λιγότερα λόγια, περισσότερες αποφάσεις βασισμένες στην πραγματικότητα της οικονομίας μας. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες που ζητούν την αλληλεγγύη των εταίρων της πρέπει να κάνει τα καθήκοντά της, πρέπει να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να μειώσει το χρέος και για να εξασφαλίσει μια ανάπτυξη. Μόνο στη βάση αυτή θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν τα κονδύλια και αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια αυτά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλα εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Για το ευρώ. Ρωτώ τον κύριο Βαν Ρομπόη. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές και θα ήθελα να έχω από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια εξήγηση. Πώς να εξηγήσω ότι το ευρώ μας αυτό το θνησιγενές, το ε, αδύναμο, πώς είναι δυνατόν να έχει μια ισοτιμία 1,40 και 40 με το δολάριο και 1,42. και 42. Αν ήταν 1 ευρώ ισότιμο με 1 δολάριο θα ήταν αρκετό. Κάνω την ερώτηση. Ε, η, λύση, όπως έλεγα, είναι περισσότερη Ευρώπη. Αυτό ισχύει και για την οικονομία μας. Και χαίρομαι που οι 27 χώρες μέλη έχουν επαναλάβει, επιβεβαιώσει και πάλι μια βασική αρχή, δηλαδή της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Δεν, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μια αφηρημένη αρχή. Αντιθέτως, είναι το κλειδί για την διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας. Η ανταγωνιστικότητά μας είναι αυτή που θα αποτελέσει την βάση για τη στρατηγική 2020. Η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που θα στηρίξει το κοινωνικό μας μοντέλο. Η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που θα στηρίξει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών μας, των μεγάλων επιχειρήσεών μας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομία, με δύο λόγια της απασχόλησης. Και έρχομαι σε ένα παράδειγμα, γιατί καλό είναι κάπου κάπου να βρίσκουμε και κανένα θετικό παράδειγμα. Η αεροπλοεία. Στο ε, αεροδρόμιο Λεμπουρζέ που γίνεται η μεγάλη ε, έκθεση. 130 νέες ε, παραγγελίες έγιναν. Να λοιπόν ένας τομέας που είναι επιτυχημένος. Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να βασίζεται και σε ένα βάθεμα της ενιαίας μας αγοράς. Μια μείωση των βαρών για τις επιχειρήσεις που συχνά είναι σημαντικές οι επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα και μια σύγκληση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών μας. Χαίρομαι για την απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουν τη δημοσιονομική πολιτική και τη σύγκρισή της πιο φιλόδοξη. Αυτό ισχύει και για τη μεταναστευτική πολιτική. Πάλι εδώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανεγνώρισαν ότι η λύση δεν μπορεί να είναι αυξημένη έλεγχη στα σύνορα. Εγώ απάντησα σε μια ερώτηση στην τηλεόραση σε ένα πρόσωπο που διέπεται απροστατευτικό πνεύμα και θέλει να προστατεύσει τους πολίτες μιας χώρας συγκεκριμένη, δεν λέω πια. Αν θέλετε να τους προστατεύσετε καλύτερα, σύμφωνοι. Αλλά για να τους προστατεύσετε καλύτερα, καλύτερα να τους δώσετε θεωρήσεις, βίζα δηλαδή, για να έρθουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι ο χώρος Σέγγεν είναι από του πιο σταθερού πυλώνε πάνω στους οποίους βασίζεται η Ένωση. Είμαι βέβαιο επίση ότι η κατάργηση των συναριακών ελέγχων πρέπει να βασίζεται και σε ένα αυξημένο μέτρο εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο ισχυρή εάν είναι πιο ενωμένη. Αυτό ζητούμε για τα 500 τόσα εκατομμύρια Ευρωπαίων. Και όπω οι φίλοι μα οι κρόατε που επιθυμούν να ενταχθούν σε λίγου μήνε και εδώ συγχαίρω τον Πρωθυπουργό τη Κροατία που κατόρθωσε η χώρα του να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονταν, καθώς επίσης και με πλήρωση όλων των κριτηρίων. Όλες και όλοι έχουμε ακόμη στη μνήμη μας τα τραγικά χρόνια των πολέμων στην Βαλκανική Χερσόνησο. Τώρα προσφέρονται προοπτικές για ένταξη σε όλες τις χώρες της περιοχής αυτής. Αυτό σημαίνει ένα πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για όλους μας αλλά και για τους λαούς των χωρών αυτών. Τελειώνοντας θα πω ότι η ομάδα του Λαϊκού Κόμματος εγκρίνει τις, ε, τα πορίσματα του Συμβουλίου για την Μεσόγειο και για τις χώρες εκείνες οι οποίες φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε έναν δρόμο δημοκρατίας αλλά και κατά εκείνων που καταπιέζουν τους λαούς τους. Την προηγούμενη Παρασκευή οι επικεφαλής των κρατών μας έπαιξαν ένα στίχημα. Προτίμησαν να ενισχύσουν, να ενθαρρύνουν τις χώρες που βρίσκονται στις δυσκολίες αντί να τις δακτυλοδεικτήσουν σε μια προσπάθεια ωστόσο απαραίτητη της εξυγίανσης των δημοσιονομικών τους. Των δημοσιονομικών όλων μας εν τέλει. Αυτή την υπεύθυνη στάση αναμένουμε, υποστηρίζουμε και αναμένουμε να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος κύριος Μάρτιν Σούλτς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε το έργο αυτής της έκτακτης, έκτακτης διάσκεψης των Προέδρων είναι να σχολιάσει όπως εσείς εκθέσατε αυτά τα οποία εκθέσατε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κύριε Πρόεδρε Φανρόμπο υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου για τα όσα έγιναν μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και αυτά τα οποία εσείς κύριε Μπαρόζο ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας εκθέσατε. Και πρέπει να σας πω το δικό μου αίσθημα που αποκόμισα εγώ μετά από τις εκθέσεις και εισηγήσεις σας και μετά από την ανάγνωση των δημοσιευμάτων αυτού του Σαββατοκύριακου και της αρχής αυτής της εβδομάδας είναι διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που άκουσα εγώ από τις εισηγήσει σας και αποκόμισα ως εντύπωση. Έχω την εντύπωση όταν σας παρακολουθώ ότι δεν έχουμε προβλήματα, ότι όλα είναι υποέλεγχο ότι κατά το μάλλον οι ήττων πάνε όλα καλά και ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων <coughs> στην Ευρώπη έχουν δώσει την ορθή κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το βλέπει κανείς έτσι βέβαια. Όμως επιτρέπω στον εαυτό μου να πω ότι εγώ έχω κάποιες άλλες εντυπώσεις, μια άλλη διαφορετική εντύπωση. Πιστεύω ότι οι συζητήσει που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα προπαρασκευάζοντα αυτό το Συμβούλιο δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε ω πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων είναι να συγκρίνουμε. Αυτό ζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά εσεί ε, ε, παρουσιάσατε και να δούμε, να τα συγκρίνουμε, να τα αξιολογήσουμε και να τα ερμηνεύσουμε. Ένα μικρό παράδειγμα. Για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα εξήγησα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τον στόχο την δημοκρατική αποτελεσματικότητα τη Ευρώπη να την ξανακερδίσει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου για το οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αποφασιστεί στο six-pack της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω αυτού του πακέτου, αλλά από τις αξιολογήσεις κάποιων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης ε, στη Νέα Υόρκη, που άλλους αξιολογούν με θετικό τρόπο και άλλους τους υποβαθμίζουν. Με ποια κριτήρια όλα αυτά για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ποιος τους δίνει αυτές τις εντολές να αξιολογούν με αυτόν τον τρόπο. Και πάντα πριν από την αρχή ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή ενός ΕΚΟΦΗΝ να ζητείτε αξιολόγηση με το συμπέρασμα όλα προς τα κάτω να αξιολογούνται. Με αποτέλεσμα οι ζητούμενες προσπάθειες εξυγίανσης στην Ελλάδα που υπάρχουν με δρακόντιες περικοπές στο δημοσιονομικό επίπεδο, στον προϋπολογισμό, να δίνουν χρήματα για τα τοκοχρεωλήσια, για την εξόφληση χρεών και μάλιστα με υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από αυτές τις, ε, ε τους οίκους αξιολόγησης. Συζήτησε αυτό το θέμα των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διαβάζω στις ότι ο Πολωνός λέει Πρωθυπουργό λέει και είναι ο επόμενο Προεδρεύων του Συμβουλίου ότι η ελευθερία ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρώπη είναι ένα εγγυημένο κεφάλαιο που η πολωνική κυβέρνηση θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Σίγουρα έχει πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Γάλλος πρόεδρος λέει πρέπει να ελέγχεται λέει η ελευθερία. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διατύπωση του Γάλλου Προέδρου. Καθένας έχει τους λόγους του για αυτά που δηλώνει βέβαια. Αλλά δεδομένης μιας συνεκτικής προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την, για μια τέτοια ερμηνεία για το Σέγγεν δεν μπορεί να κάνει κανείς λόγο. Κύριε Φανρόμποη, μας ζητήσατε ως νομοθέτες να κάνουμε κάτι περισσότερο τώρα πια. Μια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε, είπατε εσείς ολοκλήρωσε αυτά τα πράγματα για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, να εγκρίνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Δύο ερωτήσεις έχω επ' αυτού παρακαλώ. Από πότε ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ασχολείται με εξειδικευμένο νομοθετικό έργο. Αυτό είναι ουσιαστικά δουλειά του Συμβουλίου και όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά η Ουγγρική Προεδρία θα έπρεπε να είχε διαμαρτυρηθεί. Γιατί αν ερμηνεύω σωστά τη συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο καθορίζει κατευθυντήριε γραμμέ και προσανατολισμού. Τώρα ακούω ότι προφανώ έχετε εμπλακεί στην, στο εξειδικευμένο νομοθετικό έργο σε τέτοιο βαθμό που ζητείτε από εμά να εγκρίνουμε το έργο σα, λέτε. Έχω ερωτήσει, δύο ερωτήσει. Πρώτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε την τελική ψηφοφορία την προηγούμενη Πέμπτη για δύο ερωτήσει που εκκρεμούσαν. Πρώτη ερώτηση, πρώτο θέμα. Και είναι ερώτημα προ την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ τη Ομοσπονδική Γερμανία. Τι γίνεται με την ασυμμετρική σχέση όσον αφορά την μελλοντική οδηγία και το πλαίσιο για τι ε, μακροοικονομικέ ανισορροπίε, μη ισόρροπε σχέσει. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα αφορούσε τον πρόεδρο Σαρκοζή κυρίω. Επειδή εκείνο ήταν εκείνο, ο οποίο ήταν στον ισχυρότερο βαθμό κατά της αντίστροφης ε, ειδική πλειοψηφίας των δύο τρίτων για τους ε, μηχανισμούς κυρώσεων σε υπέρβαση ελλημάτων και υπερχρέωσης. Ένα από τα σημεία σε αυτό το Συμβούλιο, διότι το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα θα μπορεί να δρομολογήσει κυρώσεις και το Συμβούλιο θα μπορεί να σταματήσει μόνο με δύο τρίτα ή με δύο τρίτα θα μπορεί να δρομολογηθεί με την κύρωση είναι αποφασιστική σημασία σε ερώτημα. Τι είπε επ' αυτού το Συμβούλιο παρακαλώ. Αν και όταν μας δώσετε την απάντηση από αυτού, τότε θα μπορέσουμε να απαντήσουμε αν αυτά τα δύο θέματα για τα οποία αναβάλαμε την τελική ψηφοφορία, στην τελική ψηφοφορία που προβλέπεται για τον Ιούλιο, θα οδηγήσει στο να μπορέσει να εγκρίνει ή να απορρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό μην με παρεξηγήσετε και μην ενοχληθείτε από αυτά τα οποία λέω. Πολλά από αυτά τα μπόρεσα να τα αποκομίσω από δημοσιεύματα στον τύπο. Πολλά από αυτά τα οποία εγώ θα ήθελα να σας ε, ερωτήσω ανέμενα να τα είχα μπορέσει να τα αντλήσω από την δική σας εισήγηση. Δυστυχώς από αυτή τη διάσκεψη προέδρων δεν έμαθα πολλά περισσότερα από όσα ήξερα πιο πριν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος της ομάδας των φιλελευθέρων. Φεχόστατ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Βαν και τον κύριο Μπαρόσο για την παρουσίαση των εργασιών του Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα αφορά βέβαια την Ελλάδα και τη συζήτηση του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης. Ας το ξεκαθαρίσουμε, η κρίση συνεχίζει να σοβεί. Σήμερα το απόγευμα συζητιέται το θέμα στην Ελληνική Βουλή Σήμερα τα spread για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία πέρασαν τα 900 σημεία. Λοιπόν, οι αγορές μας κοιτάνε και το θέμα δεν, θε, είναι μόνο μια λύση για το ελληνικό πρόβλημα, αλλά μια δομική λύση συνολικά για το πρόβλημα. Με μια ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση, με ένα πιο ενισχυμένο πακέτο από αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται μόνο κυρώσει για τι χώρε που δεν φέρουν ει πέρα στι υποχρεώσει του, αλλά απαιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι τα κράτη-μέλη να είναι υπεύθυνε να κατευθύνουν και να αποφασίζουν. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Τα κράτη-μέλη δεν αυτοτιμωρούνται. Δεν το έκαναν στο παρελθόν και δεν σκοπεύουν να το κάνουν στο μέλλον. Αυτό είναι λοιπόν ο λόγο, κύριε Πρόεδρε για τον οποίο το Κοινοβούλιο επέμεινε στο, στην αντίστροφη πλειοψηφία, στο σύστημα ψηφοφορίας με αντίστροφη πλειοψηφία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις και το Συμβούλιο εκ των υστέρων ε, να αποφασίσει ίσως ότι θα την ανατρέψει αν θέλει. Νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη θέση από πλευράς Κοινοβουλίου. Μην μας λέτε ότι είμαστε ανεύθυνοι. Αυτό το πακέτο έγινε εδώ και δέκα μήνες σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον από αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Και σήμερα ο κύριος Λίψκι, το αφεντικό του Δέλτα λίγες εβδομάδες, όπως και ο κύριος Γκάιτνερ, ο Υπουργός Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και ο κύριος Τρισέ βέβαια της Κεντρικής Τράπεζας, το ίδιο λένε με το Κοινοβούλιο, ότι απαιτείται ένα ισχυρότερο πακέτο και ένα πιο τολμηρό πακέτο. Και δεν είναι και τόσο δύσκολο να έχει κανείς ένα τέτοιο πακέτο κύριε Πρόεδρε. Αρκετό είναι το να πει το Συμβούλιο ναι στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις λογικές προτάσεις τις οποίες κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πείτε ναι λοιπόν τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Όχι. Δεν είναι τόσο δύσκολο το θέμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα ναι πείτε από πλευρά σας και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το πακέτο στο Στρασβούργο. Ένα άλλο θέμα τώρα το Σέγγεν και ο κίνδυνος διάλυσης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι κατάλαβαν τη θέση του Συμβουλίου. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Από αυτά τα οποία μας είπατε δεν κατάλαβα τίποτα σχετικά με το Σέγγεν. Τι αποφασίσατε. Στα πλαίσια του κεκτημένου του Σέγγεν υπάρχει η δυνατότητα σε δύο περιπτώσεις για επανεισαγωγή εσωτερικών ελέγχων για λόγους εθνικής ασφαλείας και για λόγους ε, σοβαρού προβλήματος ένομης τάξης. Λοιπόν, δημόσιας τάξη, συγγνώμη, γιατί πρέπει να χρειάζεται και μια τρίτη περίπτωση, μια τρίτη δυνατότητα που να συνδέεται με τη μετανάστευση ειδικά. Αυτό δεν σώζει το Σέγγεν, αυτό σκοτώνει το Σέγγεν. Και θα πρέπει να το επαναλάβω και στα γαλλικά. Ίσως στα γαλλικά ε, να το καταλάβουν καλύτερα. Υπάρχει ένας λόγος λοιπόν. Το Σέγγεν δεν θα σωθεί αλλά θα δολοφονηθεί με αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου. Και μαζί με το Σέγγεν θα δολοφονηθεί και η ιδέα η βασική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει λοιπόν Πρόεδρε να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα ότι το σύνολο του Κοινοβουλίου είναι ενωμένο εδώ σε σχέση με αυτό το θέμα και δεν θα ψηφίσει μια νέα δυνατότητα επανεσαγωγής μεθοριακών ελέγχων ούτε σήμερα ούτε ποτέ. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη δεν είναι η ενίσχυση των εσωτερικών συνόρων είναι η ενίσχυση των κοινών εξωτερικών και αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι μια κοινή πολιτική για το άσυλο. 12 χρόνια την περιμένουμε. Μια κοινή μεταναστευτική πολιτική όπως το λέει και η συνθήκη άλλωστε και όπως επίσης λέει η συνθήκη πρέπει να μοιραστούμε το βάρος αν υπάρξει μια μαζική θα έλεγα εισρωή μεταναστών όπως έγινε όταν 300.000 κάτοικοι του Κωσυφοπεδίου ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνη την εποχή δεν χρειαζόμασταν μια τρίτη εξαίρεση για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Είχαμε μια μεταναστευτική πολιτική και αντιμετωπίσαμε με αλληλεγγύη το πρόβλημα. Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είμαστε στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα το επιτρέψει. Ο επόμενος ομιλητής. ECR. Uh, uh, Πριν να αναφερθώ στα θέματα αυτά, θα έρθω λίγα, λίγο σε ορισμένα από τα αυτά που είπε ο, ο κύριος Βαν Ρομποϊ, που είπε πρώτα ότι είναι ηθικά και πολιτικά απαραίτητο να προσφέρουμε υποστήριξη σε όλες τις χώρες εκείνες στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή που επιθυμούν να ε, καθιερώσουν θεμελιώδεις ελευθερίες σε κράτος δικαίου. Πρόκειται για ιστορική ευκαιρία ε, να καταφέρουμε ένα ισχυρό πλήγμα κατά των εξτρεμιστών και εδώ και στο εξωτερικό που συχνά μιλούν για σύγκρουση πολιτισμών. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά είναι μάλλον ανάμεσα στους πολιτισμένους ανθρώπους όλων των φυλών και όλων των θρησκειών και στους βαρβάρους πάλι όλων των φυλών και θρησκειών οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους με τον φόβο και τον τρόμο. Και αυτές οι συγκρούσεις για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, οικονομική ανάπτυξη για να αυξηθεί η απασχόληση και να μειωθεί η φτώχεια και τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για να αντιμετωπίσουμε ορθά εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να μας καταστρέψουν. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Αγαπητέ Ζωζεφ, εδώ δεν χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, αλλά καλύτερη Ευρώπη χρειάζεται να εφαρμοστεί καλύτερα η φυστάμενη νομοθεσία και χρειάζεται οι φυστάμενοι μηχανισμοί και οργανισμοί να είναι πιο αποτελεσματικοί. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι απέναντι σε πραγματικότητες πραγματικές, σε ε, κινδύνους πραγματικούς. Το πρόβλημα, το διαμεθοριακό πρόβλημα είναι πραγματικό. Η τρομοκρατία είναι πραγματική απειλή και η μεγάλη κλίμακα μετανάστευση αποτελεί πράγματι πρόκληση. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και αποφασιστικοί, να είμαστε δίκαιοι αλλά σταθερή, να διατηρηθούν ο έλεγχοι στα σύνορα όπου αυτή είναι απαραίτητη και ιδίω για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου όπου αυτή είναι εθνική. Και όπου δεν υπάρχουν πλέον πρέπει να αντικατασταθούν με μέτρα τα οποία θα προκαλούν εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα. Ό,τι αφορά του Ρώμα, θεωρούμε ότι ήταν σημαντικό που τέθηκε το θέμα. Η ένταξη των Ρώμα με σεβασμό των θεμελιωδών του δικαιωμάτων είναι ζήτημα συνείδηση και κάτι που ανησυχεί όλου μα. Για την Κροατία. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι προχωρούν καλά οι διαπραγματεύσεις και πλησιάζει η μέρα όπου ε, θα προσχωρήσει η χώρα αυτή. Για την οικονομική κρίση είναι σημαντικό για μας όλες οι χώρες να παίξουν πλήρως τον ρόλο τους μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Μέσα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα η Ευρωζώνη. Και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τους κανόνες της Ευρωζώνης πρέπει να είναι υπεύθυνοι και για τα ε, προβλήματά του, τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Αυτοί που παραβίασαν το σύμφωνο σταθερότητας οφείλουν τώρα να υποστούν τις συνέπειες. Και δεν είναι αληθές κύριε Βεχόφστατ που λέτε ότι ποτέ μια χώρα δεν ε, αυτοτιμωρήθηκε. Η Γερμανία είναι ένα συναρπαστικό παράδειγμα. Από τον Έρχαρτ και μετά άσκησε μια αυστηρή, μια ε, πολιτική λιτότητα αυτοτιμωρούμενη για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρομερός κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε λόγω της κρίσης στην Ευρωζώνη. Δεν αντιμετωπίσαμε όρθα την ε, υποβόσκουσα οικονομική κρίση με περιορισμένες ε, επενδύσεις, μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπονομεύει όλους μας. Χρειαζόμαστε ενίσχυση των βιομηχανιών μας. Σήμερα το μέγα θέμα ίσως είναι η Ελλάδα. Αλλά όταν θα γραφεί η ιστορία του 21ου αιώνα, το θέμα θα είναι πώς θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση για να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό αυτό παλιροϊκό κύμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρεμπέκα Χάρμς των Πρασίνων παρακαλώ. Συμπρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φανρόπα, κύριε Μπαρόζο και εσάς. Εξοργίστηκα για αυτά που είπατε για τη συνθήκη Σέγγεν και για τον ισχυρισμό ότι το Συμβούλιο λέει εργάζεται για μια βελτίωση. Μου φαίνεται κοινική αυτή η παρατήρηση. Θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά. Πώς καταλήξαμε σε αυτή τη συζήτηση. Οι Ευρωπαίοι την Αραβική Άνοιξη σχεδόν την προσπέρασαν, την έχασαν, διότι η συνεργασία με τα αυταρχικά καθεστώτα στον αραβικό κόσμο και στην Βόρεια Αφρική ήταν τόσο καλή στο παρελθόν. Τώρα διοργανώνονται στρογγυλές τράπεζες για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση. Και ταυτόχρονα μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται στεγανά και αυτά τα στεγανά στρέφονται ακριβώς κατά των ανθρώπων που έναντι πολέμου και καταπίεση στον αραβικό κόσμο αντιδρούσαν και ήθελαν να διαφύγουν. Είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη αυτή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Κύριε Φαν είναι και μάλιστα ως ο πρώτος είσαστε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς δεν μπορείτε σοβαρά να εκπροσωπείτε μια τέτοια άποψη. Ότι η κατάργηση λέει του Σέγγεν, της συνθήκης του Σέγγεν είναι βελτίωση. Αυτό θα έπρεπε να το αποσύρετε ως παρατήρηση, να ακυρώσετε αυτή σας την παρατήρηση. Ελπίζω ότι η συζήτηση θα καταδείξει τώρα σήμερα ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ό,τι μπορεί θα κάνει, ώστε να παραμείνει στην απόφαση αυτή για το Σέγγεν. Και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο εσείς εκπροσωπήσατε και είναι πολύ αντιδημοκρατικό. Σε μια τέτοια σοβαρή απόφαση να προσπαθείτε εσείς να αποκλείσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο σημείο, Ελλάδα. Δεν θα επαναλάβω κι εγώ αυτά τα οποία ακούστηκαν. Πολλά σημαντικά αναφέρθηκαν για την οικονομική διακυβέρνηση. Όμω μία πτυχή θα ήθελα να τονίσω με έμφαση σε αυτή τη συζήτηση και προσπάθησα να το κάνω την προηγούμενη εβδομάδα ήδη. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες, μια και έχουν τέτοια μορφή τα πακέτα περικοπών και λιτότητας, δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Ξέρετε, χρειαζόμαστε νέο καθορισμό των συνθήκων πλαισίου υποστήριξης για την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ένα πακέτο επενδυτικών μέτρων ώστε να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία. Τι στοχεύετε να κάνετε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση, εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, παρόλα όσα μας είπατε. Απουσιάζει εδώ απόλυτα μια σοβαρή πτυχή και αυτή είναι πολύ σημαντική, κέρια σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, δίκαια μέτρα και σε αυτή την περίοδο κρίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, διασφαλίζοντας αυτή την πτυχή για τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να ενισχυθεί και να, παροτρα... να... να ενθαρρυνθεί ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδας ε, Γιώργος Παπανδρέου να συμμετάσχουν οι πλούσιοι σε αυτή την εισφορά τη συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και οι τράπεζες. Γιατί είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και της δικαιότητας. Είμαι βαθιά πεισμένη μετά από την συζήτηση και αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή ιστορία και την ιστορία αυτής της Υπήρου ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη είναι για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Και η μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή υπόσχεση πάντα έβαινε εκ με την υπόσχεση για δικαιοσύνη, για καλύτερη ανα αναβαθμισμένη, πιο δίκαια ζωή στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα κατάφερε μέχρι σήμερα. Και μάλιστα σε αυτή την κρίση που περνάμε δεν τα κατάφερε καθόλου να τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Πιστεύω ότι η επιστροφή στα εθνικά κράτη, η επιστροφή των εθνικών κρατών καλύτερα θα μπορούσε να ε, είχε λειτουργήσει αν ε, οι Ευρωπαίοι είχαν ε, εκφραστεί υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης με καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Αριστεράς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, ο κύριος Λόταρ Μπίσκι. Θυμάμαι ότι ο κύριος Μάρτιν Σούλτς για αυτή την διάσκεψη κορυφής μίλησε για μια ιστορική σημασία σύνοδο κορυφής για το μέλλον της Ευρώπης. Όμως δεν υλοποίησε πιστεύω αυτή η σύνοδος κορυφής την υπόσχεση αυτή. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για τα πακέτα και τα μέτρα για την οικονομική διακυβέρνηση ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 2020 απασχόληση, ενεργειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση δεν ήταν δυνατόν ούτε στην Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων να επιτευχθεί μια συμφωνία. Πόρο απέχει μια συμφωνία για το πρόβλημα της Ελλάδας. Μια ματιά στο σημερινό ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες της Ευρώπης δεν πιστεύουν ότι σύντομα θα βρεθεί η σωστή πορεία για να διαφύγουμε από αυτή την κρίση. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά επειδή συνεχίζουμε να παραμένουμε πιστοί στην ίδια οικονομική πολιτική που μας οδήγησε σε αυτή την κρίση στο παρελθόν. Και απαιτείται από την Ελλάδα να εγκαταλείψει την θεμητή δημοκρατική της πολιτική να καταργηθούν νομοθετήματα και να υπάρξει η περικοπή, η περιστολή δαπανών και μόνο τότε θα υπάρξουν πιστώσεις δάνεια που θα δοθούν στην Ελλάδα και μάλιστα σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δείχνουν όλα αυτά ότι αυτή η θεραπεία μορφής σοκ γίνεται κανόνας, θα μπορούσε να γίνει κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία πολλά έχουν μάθει και μπορούν να μας πούν για αυτή την ιστορία. Και βλέπουμε ότι υπάρχει απειλή ιδιαίτερα έντονων κυρώσεων όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Εδώ μία εσφαλμένη οικονομική διακυβέρνηση βρίσκεται υπό εξέλιξη για, τις, ε, για τους οίκους ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης ακόμα περισσότερο καθορίζουν σήμερα αυτές οι δράσεις τους με ποιους κανόνες παίζεται το παιχνίδι. Η, Ευρωπαϊκή, όμως, ε, Ευρωπαϊκή, η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όμως στο περιθώριο. Οι Έλληνες σήμερα και αύριο έχουν, απεργούν και μάλιστα μαζικά. Και κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Βουλή των Ελλήνων αύριο απορρίψει το μεσοπρόθεσμο, τη μεσοπρόθεσμη συμφωνία. Μπορείτε να πείτε είναι θεωρητικό αυτό το ερώτημα, ίσως, αλλά διαρωτώ με γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα Β ή πρόγραμμα Γ, αναδίπλωσης Β ή Γ για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο δεν θέλουμε να συμβεί, αλλά αν συνέβαινε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ ο κύριος Νάιζελ Φάραντς, Ελευθερία και Δημοκρατία. Α, ωραία, έχουμε όλους τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μπροστά μας που μας λένε ότι όλα είναι μια χαρά. Ναι, ναι, ωραία, θα το κεφάλι σας στην άμμο, αλλά οι υπόλοιποι μας κοιτούν. Η Ευρώπη ζει με δανεισμένο χρόνο, με δανεισμένα χρήματα. Αυτή η δεύτερη διάσωση της Ελλάδας στην ουσία παρατείνει την αγωνία της. Ό,τι και να αγορέσουν οι Κινέζοι, όσα, όσα ομόλογα μοριακά δάνεια και να αγοράσουν οι Κινέζοι, ό,τι και να λεφτά και να στείλει ο Σαρκοζή. Το γεγονό είναι ότι η Ελλάδα πτωχεύει. Δεν μπορεί να, ε, να ε, κάνει ούτε καν τι απαραίτητε δαπάνε από τον προπολογισμό τη. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτε και το όλο και πιο αποκρουστικό Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είναι να βαθαίνουν την κρίση. Υπάρχει απόλυτη απώλεια πίστη σε εσά διότι είσαστε πολιτικά ανέντιμοι. Ο τρόπος με τον οποίο περάσατε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ο δικός σας διορισμός στους Προέδρους της Ευρώπης, όλα αυτά ήταν στην πραγματικότητα απάτη. Τώρα οι άνθρωποι στην Ευρώπη πιστεύουν όχι μόνο ότι δεν είσαστε ε, έντιμοι, αλλά έρχεστε και ρυθμίζετε τα, τη ζωή τους οδηγώντας το πλοίο της Ευρώπης στα βράχια τρέχετε από εδώ και από εκεί σαν αποκεφαλισμένα κοτόπουλα. Δεν προσφέρετε σε κανέναν εμπιστοσύνη. Δεν δείχνετε ηγετική ικανότητα. Όποια πρόγνωση και να έχετε κάνει στι συναντήσει σα αυτέ, αποδείχθηκε των υστέρων ήταν εσφαλμένη. Τώρα είσαστε η συμμορία των Βρυξελών και είσαστε διαρκώ σε άρνηση να δεχθείτε οποιοδήποτε plan B, οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή, ενώ εκατομμύρια χάνουν τις δουλειές τους, φτωχαίνουν διαρκώς και στην πραγματικότητα αυτό που κάνετε είναι εγκατάλειψη καθήκοντος. Δεν είστε ικανοί. Και η παρούσα αίθουσα που ίσως είναι άδεια σήμερα διότι οι ευρωβουλευτές δεν δίνουν δεκάρα για το τι γίνεται εδώ αλλά έξω υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις που συγκεντρώνονται. Και αν απορρίψουν τις απαιτήσει σας, αν πούν όχι στο ε, πακέτο, εάν υπάρξει τελικά πτώχευση, θα είναι οδυνηρό για τις τράπεζες, θα είναι οδυνηρό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά καλύτερα έτσι παρά να παρατείνετε η αγωνία. Έχετε κανένα σχέδιο γι' αυτό. Αν δεχθούν ωστόσο τις απαιτήσει σα, μην νομίζετε ότι η, η αραβική ε, άνοιξη δεν μπορεί να γίνει ένα μεσογειακό θέρος δυσαρέσκειας και αγανάκτησης. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο αντιπρόεδρος Φίλιπ Κλάις. Μη εγγεγραμμένος. Παρακαλώ κύριε Σούλτς, σταματήστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο, λέει ο κύριος Κλάις. Πράγματι ακούστηκαν κάποια μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν το Σέγγεν να γίνει πιο αποτελεσματικό ο τρόπος όμως με τον οποίο διατυπώθηκαν τα μέτρα αυτά δεν είναι θα έλεγα ο καλύτερος. Μια ολόκληρη θα έλεγα γκάμα σταδιακά εφαρμοζόμενων μέτρων προβλέπεται και στο τέλος μόνο υπάρχει μια καταληκτική ρήτρα η οποία κατ' εξαίρεση να επιτρέπει την αποκατάσταση των, εξωτερικών, των εσωτερικών συγγνώμη, ελέγχων. Λέγει η πρόταση ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται επί τη βάση εξειδικευμένων και αντικειμενικών κριτηρίων. Με άλλα λόγια κύριε Πρόεδρε, τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να αποκαταστήσουν τους εσωτερικούς ελέγχους στην ουσία θα πνιγούν από μια διαδικαστική χιονοστιβάδα γραφειοκρατίας και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο και προφανώς δεν θα επιτραπεί η ενίσχυση των εσωτερικών σύνορων. Για τα εξωτερικά σύνορα πολλοί λέγουν για την αποτελεσματικότητα της Frontex. Χρόνια το συζητάμε αυτό κύριε Πρόεδρε και από ό,τι φαίνεται δεν ακούμε καινούριε ιδέες που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Μιλάμε και για τις εταιρικέ σχέσεις με τρίτες χώρες. Τι σημαίνει μια τέτοια εταιρική σχέση. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα μέχρι τώρα αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να μπορούν να παρέμβουν μόνες τους για να παρεμποδίσουμε έτσι την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Όχι βέβαια. Ο κύριος Μπαρόζο για μια ακόμη φορά από ό,τι ακούσαμε κατηγόρησε τους λαϊκιστές, τους εξτρεμιστές οι οποίοι θέλουν να καταστήσουν ανέφικτη την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Αντιστρέφεται την πραγματικότητα κύριε Μπαρόσο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή και όχι το Συμβούλιο η οποία απειλεί την ύπαρξη του Σέγγεν γιατί δεν εφαρμόζεται παρά το ίμιση της συμφωνίας του Σέγγεν λόγω της μη ύπαρξης ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Προφανώς ότι τα εσωτερικά σύνορα είναι διάτρητα. Αυτό δεν υπάρχει ε, αμφιβολία και αυτό προκαλεί μια απόλυτα δικαιολογημένη δυσφορία στους Ευρωπαίους πολίτες. Δείτε παρακαλώ την πραγματικότητα και προσπαθήστε να πάρετε τα σωστά μέτρα και να μας διαβάζετε τέτοιου είδους συμπεράσματα χωρίς νόημα. Διαδικασία Κατσιάη. Ε, Madame Ildiko σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πρόεδρο και θα ήθελα να συγχαρώ για να... διότι ήταν μια μεγάλη πρόκληση η Σύνοδος Κορυφής ε, και ήταν μεγάλο επίτευγμα. Τα γεγονότα μιλούν αφ' αυτόν. Έχουμε μια στρατηγική για πρώτη φορά για τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια στρατηγική για τη λεκάνη του Δούναβη και για την ε, διεύρυνση. Έχουν γίνει πολλά και σε σχέση με το έργο που έχει επιτελεστεί και από την Ουγγρική Προεδρία που είναι τόσο σημαντικό. Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν σε σχέση με οικονομικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλωσε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα και δεν αντέδρασε σωστά όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και ε, δημοσιονομικά προβλήματα που απέρευσαν από την κρίση. Και δυστυχώς δεν υπήρξε ιεράρχηση προτεραιοτήτων που να είναι σαφής για τα θέματα τα δημοσιονομικά και τα φορολογικά. Τώρα όμως βρίσκονται σε ε, ε, ορατή απόσταση ευδιάκριτα και θέλω να σας παρακαλέσω να γίνουν τα αναγκαία μέτρα, να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Όπως είπατε, το τέλειο, το καλύτερο δεν πρέπει να είναι ο εχθρός του καλού. Ευχαριστώ. Όλα αυτά δείχνουν την τάση που υπάρχουν στις οικονομίες μας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο βήμα, ένα μεγάλο μάθημα ότι η λιτότητα μόνη της δεν λειτουργεί. Το αντίθετο, όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτή η συνταγή, όπως δείχνει η ελληνική οικονομία, η πορτογαλική, η ιρλανδική, ήταν λανθασμένη σε σχέση με τις αγορές. Αναμένω το Συμβούλιο να υιοθετήσει μέτρα ευρωπαϊκά αλληλεγγύης, όπως τα ευρωομόλογα, για την αντιμετώπιση του εθνικού χρέους. Να υπάρξει φόρος τέλος στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να προχωρήσουμε στη συνεργασία την οικονομική και την πολιτική όσον αφορά τις εμπορικές μας σχέσεις ώστε να υπάρξει η σωστή ισορροπία στη συνεργασία αυτή μεταξύ των κρατών μελών. Αναμένω το Συμβούλιο να ε, υποχρεώσει σε σχέση με τις τράπεζες ε, να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των φορολογικών παραδείσων ε, όσον αφορά τα κονδύλια που χρειάζονται. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σε σχέση με το, με το πρόγραμμα του Συμβουλίου. Αν κάτι πάει στραβά, ποιο είναι το πρόγραμμα Β αναδίπλωσης σε σχέση με την νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται εις βάρος των πολιτών. Αυτό όχι μόνο υπερχρεώνει την Ελλάδα και επιδεινώνει την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, Γκραμ Βότσον, παρακαλώ. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις για τη μείωση ουσιαστικά του κοινωνικού κεκτημένου, του κοινοτικού κεκτημένου, μέσω της επανεισαγωγής των εσωτερικών μεθοριακών ελέγχων. Νομίζω ότι σκοπεύει να διαφοροποιηθεί με τέτοιο τρόπο το Συμβούλιο από τις κινήσεις των λαϊκιστών στο μέλλον και πώς θα εξηγήσει στους ιστορικούς ο κύριος Βαν Ρόμπαϊ ότι αυτό το οποίο είπατε σήμερα ότι είναι κατόρθωμα ευρωπαϊκό στην ουσία έγινε από τη δική σας Προεδρία δυστυχώς. Εσείς τελικά τι θέλετε να παίξετε το βρούτο στον κάσιο του Συμβουλίου σε ένα πράγματι απέσιο λαϊκιστικό θέαμα. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε πρόεδρε Φαν αντιμετωπίσατε ε, μία από τις πιο περίπλοκες ημερήσιες διατάξεις στο τελευταίο συμβούλιο στο οποίο πήρατε από τότε που είστε πρόεδρος. Και πράγματι αμφισβητείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά θέματα πλέον. Παρ' όλα αυτά σημειώθηκε πρόοδος, αν και πολλοί δεν την αναγνωρίζουν, κάποιοι από τους συναδέλφους μου. Υπήρξε πρόοδος σε σημαντικούς τομείς. Θα ήθελα εγώ να υπογραμμίσω το πού βρισκόμαστε σχετικά με το πακέτο διακυβέρνησης, οικονομικής διακυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται, όλη η προσοχή στρέφεται σε μια πολύ περίπλοκη λύση την οποία θα πρέπει να βρούμε για την ελληνική κρίση του ευρώ, λέει η ομιλήτρια. Το θέμα δεν είναι η πυρόσβεση όμως κύριε Πρόεδρε. Η πυρόσβεση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πακέτο προτάσεων για την αποτροπή αντιστοίχων κρίσεων στο μέλλον που θα διασφαλίσει την ανάπτυξη ε, και ε, την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είμαστε σύμφωνοι κατά 98%. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της συμφωνίας. Απευθύνατε έκκληση λοιπόν προς εμάς και εμείς απευθύνουμε έκκληση προς εσάς στο Συμβούλιο. Η κυρία Γιακονσάρη, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθένας από μας μπορεί την σημερινή οικονομική κρίση να τη συγκρίνει με έναν παγκόσμιο πόλεμο χωρίς ε, διακήρυξη πολέμου και ταυτόχρονα έχουμε τεράστια υπερχρέωση των ΗΠΑ. Γνωρίζουμε ότι ο ρόλος της Κίνας είναι δεδομένος σε αυτό το πρόβλημα. Πρόκειται για πολύ σοβαρά βαθιά προβλήματα και είναι ανθρώπινο, απόλυτα ανθρώπινο. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Φαν Ρόμπαϊ, αυτό που είπε δεν ήταν μια συνήθις ε, συνεδρίαση και η ίδια η κατάσταση δεν είναι συνηθισμένη κατάσταση και γι' αυτό η σύνοδος αυτή δεν μπορούσε να είναι μια συνήθις σύνοδος. Όμως η συζήτηση αυτή νομίζω ιδιαίτερα και έντονα διαρθρώνεται και επικεντρώνεται μέσω του ότι ο λόγος σας ιδιαίτερα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο και δεν με καθησύχασε καθόλου. Το ερώτημα είναι, το ζήτημα είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Έχει ένα πραγματικό αυθεντικό πρόγραμμα. Πώς δηλαδή και τι θα γίνει ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε μια ε, εμβάθυνση και ένα βάθεμα και μια πιο δυνηρή μορφή της κρίσης. Πολλά διάβασα και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά κάτι να κάνουμε ώστε να μην γίνει πιο βαθιά η κρίση. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε ήδη, σήμερα και αύριο στην Ελληνική Βουλή συζητείται και θα τεθεί για ψηφοφορία ένα νέο πρόγραμμα σκληρής λιτότητας και ιδιωτικοποίησεων. Ο κόσμος είναι στους δρόμους. Κύριε Ρομπάη και κύριε Μπαρόζο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση γίνεται κάτω από την απειλή. Αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν θα πάρει η Ελλάδα την πέμπτη δόση του δανείου δεν θα συζητηθεί το θέμα της νέας οικονομικής βοήθειας. Θα ήθελα σας παρακαλώ, επειδή είναι κρίσιμες οι στιγμές, να θέσω με μεγαλύτερη ενδεχομένως σαφήνεια το ερώτημα που ήδη σας ετέθη. Στην περίπτωση που δεν ψηφιστεί το νέο πρόγραμμα λιτότητας, θα πραγματοποιήσετε την απειλή, δεν θα δοθεί η πέμπτη δόση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πέρα από τις επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνική πραγματικότητα, υπάρχει πρόβλημα για την Ευρωζώνη. Έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο θα παρακαλούσα σαφή απάντηση γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές και οικονομικά και πολιτικά όχι μόνο για την ελλάδα αλλά και για την ευρώπη. Ευχαριστούμε το Συμβουλίο για την παρουσία του εδώ και τον Πρόεδρο Μπαρόσο της Επιτροπής. Λυπάμαι που οι διασκέψεις μας γίνονται με αυτή τη μορφή και διαρωτώ αν είναι συμβατές με το άρθρο 15 της Συνθήκης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε, είναι μια επιπλέον συνθήκη αυτό το πράγμα. Το μια συνθήκη η οποία δεν έχει κοινοτική διάσταση ουσιαστικά. Διαρωτώ με πώς τα πλαίσια αυτού του μηχανισμού που εμπλέκει πάρα πολύ ψηλά ποσά να προβλέψουμε τον κοινοβουλευτικό και πολιτικό έλεγχο. Το ελεγκτικό συνέδριο θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο. Τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ποιος θα ασκεί τον πολιτικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο θέματα. Πρώτο, για τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με το σύμφωνο το πακέτρο έξι νομικών κειμένων και κάνω λόγο ως εισηγήτρια για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι ένα απόλυτα νέο Αυτό όμως το οποίο πρέπει να αποφασιστεί και είναι τεράστια σημασία είναι μέσα στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης που χρησιμοποιήθηκε από όλους που παρενέβησαν ε, την ε, ημέρα αυτή στο κείμενο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και που αποκλεί το Συμβούλιο οποιαδήποτε δυνατότητα να εξεταστούν σοβαρά τα πλεονάσματα ταυτόχρονα όμως ενώ αξιολογούνται τα ελλείμματα. Σε ένα θέμα αλληλεξάρτησης δεν μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα στις χώρες που έχουν ελλείμματα χωρίς να προσέξουμε ότι αυτό συνδέεται ιδιαίτερα με τα πλεονάσματα άλλων χωρών υπάρχει αλληλεξάρτηση. Η πολιτική θέση του Συμβουλίου να αποκλειστεί αυτό το, αυτή η πλευρά των προβλημάτων σε σχέση με τις ανισορροπίες δεν είναι σωστή. Τι γίνεται εδώ προς την Επιτροπή δεύτερον. Είναι σημαντική ανάπτυξη. Χωρίς την ανάπτυξη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ήθελα να πω μόνο δύο πέρασε ο χρόνος σας. Ελαστικότητα λέει η ομιλήτρια και να υπάρξει απλούστευση γραφειοκρατική, ανακούφιση γραφειοκρατική. Έληξε ο χρόνος σας κύριε, λέει ο πρόεδρος. κύριο παρακαλώ. Uh, thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί εδώ, είναι καινή αίθουσα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, πολίτες στην Ελλάδα που έχουν βγει στους δρόμους. Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να διαλύσει αυτές τις διαδηλώσεις. Και αυτή η κατάσταση είναι το δικό σας δημιούργημα, εσείς το γεννήσατε. Η Ευρωζώνη αποτυγχάνει, καταστρέφεται, είναι αλήθεια αυτό, ξυπνήστε να το καταλάβετε αυτό. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να διαλέξει είτε να επιστρέψει στη γραχμή, ίσως να είναι και ο καλύτερος δρόμος ή κάτι άλλο. Ας ακούσουμε το λαό λοιπόν. Ο λαός αποφασίζει. Εμείς οι πολιτικοί εφαρμόζουμε αυτές τις ε, αποφάσεις του λαού. Ε, τώρα λοιπόν δεν ακούμε το λαό, δεν αφήνουμε το λαό να αποφασίσει. Κύριε Βαν Ρομπάι, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτησή μας. Είχα ρωτήσει στο παρελθόν αν υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Εάν πράγματι υπάρξει χρεοκοπήσει πλήρως η ελληνική κυβέρνηση, ποια είναι η εναλλακτική λύση. Childers. Um, I will be brief because you'll notice that uh, the MEPs from Ireland, Greece and Portugal can't wait. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να χάνουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας με λόγια κενά όσοι ιδιαίτερα είμαστε από Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Έχετε ένα πρόγραμμα. Έπρεπε να το κρατήσετε μυστικό το πρόγραμμα αυτό για διάφορους λόγους. Ή μήπως δεν έχετε κανένα πρόγραμμα και πάλι ούτε και αυτό φυσικά το φανερώνετε ή από την άλλη υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να συμφέρει κάποιες χώρες μέλη και όχι κάποιες άλλες χώρες μέλη. πέτω, δεν θα απαντήσετε σε αυτά τα οποία λέω αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ευρωβουλευτές από τις χώρες αυτές δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν την κατάσταση και τις θέσεις σας. Θα θέλαμε να μπορούμε να το κάνουμε. Η κυρία Γιαννάκου παρακαλώ. Μικρόφωνο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Συμβουλίου καθώς και τον ε, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ σήμερα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ε, κύριε Πρόεδρε, η υπόθεση της κρίσης του ευρώ που με πιο έντονο τρόπο εμφανίζεται σε χώρες όπως η δική μου χώρα η Ελλάδα χρειάζεται βέβαια μια αντιμετώπιση μέτρων αμέσου αποδόσεως αλλά κυρίως χρειάζεται μια διαχρονική στρατηγική και είναι φανερό ότι ο τρόπος που έχει επιλεγεί δεν είναι ίσως ο πλέον επιτυχής. ωστόσο θα έλεγα ότι πρέπει να κληθούν οι κυβερνήσεις οι οποίες συνομολόγησαν ένα μεμοράντουμ να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. εφόσον το πρόγραμμα αυτό δεν εφαρμόζεται επιτυχώς υπάρχει plan b γιατί βεβαίως η χώρα μου και οι πολίτες της δεν έχουν καμία διάθεση να επιστρέψουν στη δραχμή. Η κυρία Ποδήματα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα δύο θέματα που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η κρίση του ευρώ και η συνθήκη Σέγγεν, βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το γεγονός ότι και τα δύο σήμερα βρίσκονται υπό απειλή, κινδυνεύουν, νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να αναζητούμε λύσεις πυροσβεστικές αποσπασματικές ότι χρειαζόμαστε λύσεις προληπτικές συνολικές και προπάντων ευρωπαϊκές. για την ελλάδα σωστά είπατε κύριε πρόεδρε ότι συζητούμε αυτή την περίοδο αυτές τις μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σταθεροποίησης ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ σε, ύψος, σε βάθος τετραετίας και θα εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα από το ελληνικό κοινοβούλιο γιατί αυτή είναι η ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος που έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη και έχει απόλυτη συνέστηση της κρισιμότητας των στιγμών. όμως κύριε πρόεδρε χρειάζονται και άλλα μέτρα για την ανάπτυξη εκτός από τη δημοσιονομική προσαρμογή και χρειαζόμαστε επίσης μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της εκροής κεφαλαίων σε φορολογικούς ε, παραδείσους εντός ο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ και τους δύο Πρόεδρους ε, σχετικά με την ενημέρωση για τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις της Συνόδου για την οικονομία της Ευρώπης γενικότερα και ειδικότερα για το πρόβλημα της Ελλάδας το οποίο με αφορά ιδιαίτερα σαν Έλληνα Ευρωβουλευτή. Αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικά, γιατί μιλάμε πολιτικά εδώ, δεν θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για την ύπαρξη κάποιου σχεδίου β όταν σήμερα το βράδυ ψηφίζεται στην ελλάδα το πακέτο των μέτρων και δεν θα ήταν δυνατόν να προλάβετε εσείς το τι θα γίνει στην ελλάδα. όμως επιπλέον θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί υποθέτω ότι μελετήθηκε και εκτιμήθηκε η διεθνής οικονομική κατάσταση η κατάσταση της ηπα στην κίνα και οι επιδράσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία στο άμεσο μέλλον οι τυχόν συναλλαγματικές ανατροπές και γενικά το πού πάει η οικονομία της ανθρωπότητος. Τι μπορείτε να μας πείτε από αυτού. Κύριε Πρόεδρε, σας υπενθυμίζω ότι το κεκτημένο Σέγγιν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ε, συνθήκης το άρθρο 77 απαγορεύει οποιαδήποτε, οποιουσδήποτε ελέγχους προσώπων που διαβαίνουν τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, οποιασδήποτε εθνικότητα και είναι τα πρόσωπα αυτά. 77 και 78.3 που απαγορεύει ελέγχους σε πρόσωπα που διαβαίνουν τα σύνορα μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Σαρκοζή, όταν μιλεί για αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, θέλει να μεταρρυθμίσει την συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απλή διακυβερνητική συμφωνία και η ρήτρα προφύλαξης που υπάρχει ήδη μέσα στην συνθήκη θα επιτρέψει σύμφωνα με τον κύριο Σαρκοζή την, τον έλεγχο της ελευθερίας διακίνησης. 1.200.000 πρόσωπα που διαβαίνουν τα σύνορα του Σένγεν θα τα ελέγχει η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε συνείδηση του γεγονότος ότι αποδυναμώνοντας το Σένγκεν αποδυναμώνεται το ευρώ το οποίο θεωρήθηκε ως ένα βήμα προς μια πιο στενή, πιο σφιχτή ολοκλήρωση. Αυτοί που στρέφονται κατά του Σέγγεν στην ουσία ροκανίζουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται το ευρώ. Το ερώτημα δεν είναι της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι τα σύνορά μας. Η εποπτεία των κινήσεων κεφαλαίου. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων όπως αυτή εφαρμόζεται σήμερα και όπως με την εποπτεία που δέχεται σήμερα πρέπει να είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων και όχι στο συμφέρον των κερδοσκόπων και των αγορών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, παρακαλώ. Παρακαλώ, λάβετε το λόγο. Τα πιο σημαντικά θέματα ήταν το Σέγγεν και η ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της Ελλάδας. Σύντομα και ανοιχτά να απευθυνθώ σε αναστραφώ σε αυτά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα συμμερίζομαι το μέλημα το οποίο εκφράστηκε τόσο ξεκάθαρα για την ελευθερία κυκλοφορίας. Να προστατευτεί το Σέγγεν και το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την ελευθερία της κυκλοφορίας και νομίζω ότι αναγνωρίζετε ότι Κανείς δεν έχει πιο έντονες απόψεις υπέρ αυτών των δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με κάθε συνέπεια ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζαμε αυτό το δικαίωμα. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις αμφισβήτησης της ελευθερίας της κυκλοφορίας και της αρχής της μη αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Όμως άμεσα, με ιδιαίτερο σθένος και επανειλημμένα κιόλας, υπήρξαν περιπτώσεις από όταν πρότειναν κάποιες κυβερνήσεις ότι δεν θα είχαν αυτές τις αρχές ως προτεραιότητά τους, αντιδράσαμε άμεσα. Και ήταν πάντα σαφής η τοποθέτησή μας, ε, χωρίς οποιαδήποτε, ε, οποιουσδήποτε δισταγμούς. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ένα πρόβλημα ανταπόκριση σε μια κατάσταση όπου τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να σεβαστούν τις δικές τους υποχρεώσεις εναντί του Σέγγεν και σε σχέση με συγκεκριμένα κράτη-μέλη όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ελέγχων των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Διότι συμφωνώ με όλους εκείνους που είπαν ότι αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι η δημιουργία νέων δυσχεριών στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ακριβώς να διασφαλίσουμε τον σεβασμό των συνόρων μας. Διότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς των πολιτών και από πλευράς των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, τότε μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε πραγματικά προβλήματα να υπάρξει το κοινοτικό και εκτιμένο και να είναι σεβαστό σε αυτά τα κράτη. Γι' αυτό θα υποβληθεί πρόταση από πλευρά μα το Σεπτέμβριο σχετικά και πιστεύω ότι η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ήταν πολύ χρήσιμη και επικοδομητική σε σχέση με αυτό και δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες των συζητήσεων, των διαβουλεύσεων, αλλά πολύ ενδιαφέροντα θέματα και παρεμβάσεις έγιναν. Και το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ θετική, θα έλεγα. Το συμπέρασμα είναι πολύ θετικό. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να ενταχθούν όλα αυτά, αντί να μείνουν εκτός να τεθούν σε μια ε, κοινοτική προοπτική, αντί να δρουν μονομερό στα κράτη-μέλη, να εισαχθεί ε, για την εισαγωγή εσωτερικών συνόρων προσπαθούμε να έχουμε μια συστημική προσέγγιση όσον αφορά τα προβλήματα αυτά για μια κοινή αξιολόγηση που θα υπάρξει για ένα πολύ στενό φάσμα και πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο για αυτή, για αυτή την υιοθέτηση μέτρων όσον αφορά τους ελέγχους και για την αξιολόγηση αυτή από πλευρά συστήματος θα είναι μέρος αυτών των διαδικασιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εμπλέκεται και θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα σε σχέση με κάτι τέτοιο είναι και σε σχέση σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, να αποφύγουμε μονομερείς αποφάσεις και εξελίξεις, διότι όπως αναφέρθηκε τα κράτη-μέλη μπορούν να εισαγάγουν περιορισμούς όσον αφορά τα εσωτερικά σύνορα. Μπορούν να το κάνουν. Το θέμα είναι, θα το κάνουν αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπως το έχουμε τώρα ή θα υπάρξει ένα πολύ πιο εξειδικευμένο πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για να γίνεται αυτό υπό ευρωπαϊκό πρίσμα. Και πιστεύω ότι είναι μια μέθοδος ενίσχυσης του κοινοτικού μας κεκτημένου και της κοινή μας προσέγγισης. Ας αναμείνετε λοιπόν, ας περιμένετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχετε την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη συζητήσετε διεξοδικά. Και αυτό θα γίνει και θα διασφαλιστεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το μεγάλο κεκτημένο για την ελευθερία κυκλοφορία των πολιτών μα και όχι μόνο πολιτών, αλλά οι ελευθερίες κυκλοφορίας που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωσή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στον σεβασμό αυτών των τεσσάρων ελευθεριών όπως γνωρίζετε και θα παραμείνει πιστή σε αυτή την αρχή χωρίς κανένα δισταγμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο ζήτημα είναι ένα πολύ ακαθόδε, πολύ δύσκολο ζήτημα για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες. Όπως πρώτα είπα πιο πριν, εξετάζουμε και για την Ελλάδα να είμαστε σαφέστεροι όσον αφορά την ανάγκη για ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη. Κατανοούμε τα μελήματα και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Κατανοούμε την απογοήτευση πάρα πολλών πολιτών, Ελλήνων πολιτών που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου φτωχαίνουν καθημερινά ενώ βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι Έλληνες παίρνουν τα χρήματά τους και τα περνάνε στο εξωτερικό και έτσι λείπουν από την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί με τους Έλληνες και με τους εαυτούς μας πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφορετικός από αυτές τις επώδυνες πολιτικές λιτότητας και περικοπών και της αναθεώρησης δημοσιονομικά ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την Ελλάδα να υπάρξει δυνατότητα ανάκαμψης και ανάπτυξης. Και αυτοί που κάνουν λόγο για ένα πρόγραμμα αναδίπλωσης, σχέδιο αναδίπλωσης Β, οι δράσεις, πρόγραμμα Β, για μια εναλλακτική άλλη λύση. Λένε ψέματα, ψεύδονται. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα Β για να αποφευθεί, να αποφευθεί η πτώχευση ή η χρεοκοπία. Το μόνο εναλλακτικό, η μόνη δυνατότητα είναι αυτή που υπάρχει τώρα ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νομισματικό την ευρωπαικη ενωση απο το διεθνε νομισματικο ταμειο με την υποστήριξη όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιοδήποτε πρότεινε ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση θα είναι υπεύθυνο για πραγματικά ολέθριε επιπτώσει όσον αφορά τα δημοσιονομικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το σχέδιο που έχουμε. Και φυσικά σχολιαστέ μπορούν πάντα να εικάζουν και να υπάρχουν υποθέσει ή να ε, ε, εικάζουν κάτι. Εδώ δεν εικάζουμε ούτε κάνουμε οικοτολογίε. Έχουμε ένα τελικό πρόγραμμα και πρέπει να τηρηθεί, να παραμείνουμε πιστό. Αυτό είναι το πρόγραμμα που υπάρχει το σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα και οποιαδήποτε προσπάθεια να υπάρχει λέει μια άλλη εναλλακτική λύση και να αμφισβητηθεί αυτό το πρόγραμμα δεν θα ενισχύσει, δεν θα τονώσει την εμπιστοσύνη για την Ελλάδα των Ελλήνων και την ε, αυτοπεποίθηση σε αυτό το πρόγραμμα. Το μήνυμα, αν θέλετε να βοηθήσετε, είναι α παραμείνουμε πιστοί και σεβαστούμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα υπάρξουν θαύματα, δεν θα γίνουν θαύματα. Δεν υπάρχουν με τη μαγική ράβδο, με το μαγικό ραβδί εναλλακτικέ λύσει στι επώδυνε μεταρρυθμίσει ε, και περικοπές και δεν θα πρέπει εδώ να αγνοήσουμε αυτή την πτυχή και όταν ζητήσετε από κάποιους ε, να δώσουν, να επενδύσουν άλλα περισσότερα κονδύλια θα πούν ούτε δεκάρα παραπάνω πρέπει να τηρηθούν αυτοί οι όροι πρέπει απόλυτα να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις φυσικά του, ε, της Βουλής των Ελλήνων του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά χρειαζόμαστε ευθύνη και αλληλεγγύη σε σχέση με την Ελλάδα μια χώρα δεν μπορεί να ζει πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες της επί μεγάλο χρονικό διάστημα διάστημα. Μια χώρα η οποία έκανε κατάχρηση αυτών των δυνατοτήτων που είχε δεν υλοποιεί τι ευθύνε τη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λοιπόν μια κοινή ευθύνη όλων μα να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με του Έλληνε εταίρου μα υπό την προπόθεση ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα στο ε, πλαίσιο του ευρώ και ομόνιμα λοιπόν, ομόφωνα αυτέ οι αποφασίσει να γίνουν σεβαστέ. Υποστηρίζονται απόλυτα από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και όταν θα έρθει η ώρα της αλήθειας ελπίζω ότι η Ελλάδα θα επιλέξει την σωστή και μόνη πορεία να διέλθει, να εξέλθει από αυτή την κρίση. Επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν θαύματα. Χρειάζονται θαραλέ, επώδυνε αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ξεπεράσει τις σημερινές τη δυσκολίες η Ελλάδα. Αν το κάνει θα έχει την απόλυτη υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Χέρμαν Φαν Ρομπάι έχει πλέον το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχάς για την Ελλάδα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία προείπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμα και χωρίς την Ελλάδα, χωρίς την Ευρώπη, συγγνώμη, η Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά της και τη δημοσιονομική της ισορροπία. Αυτό το οποίο κάνει η Ευρώπη είναι να βοηθά με δάνεια τα οποία αμφισβητούνται πολλές φορές σε διάφορες χώρες. Βοηθάει η Ευρώπη όμως έτσι ώστε η συγκεκριμένη χώρα να έχει χρόνο και να φέρει πέρα στο πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται στην πηγή του προβλήματος. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εδώ και δέκα χρόνια με έλλειψη εποπτείας, με κακές πολιτικές, αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και χωρίς την Ευρώπη υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα, υπήρχε δημοσιονομικό πρόβλημα και υπήρχε και σοβαρότατο πρόβλημα οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη είναι εδώ λοιπόν για να βοηθά έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες της χώρας και να μπει στον δρόμο της ανάπτυξης η χώρα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα σκληρότατο πρόγραμμα. Όσοι ακολούθησαν πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης στις χώρες τους και εγώ είμαι ένας από αυτούς ξέρουν ότι οι πολιτικές αυτές είναι σκληρές και καθόλου δημοφιλείς και χαιρετίζω το θάρρος της ελληνικής κυβέρνησης που αναλαμβάνει τις ευθύνε της απέναντι σε αυτές τις τρομερές εντάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Τα μέτρα αυτά και το έχουμε πει επανειλημμένα, πρέπει να είναι μέτρα τα οποία να δημιουργούν ένα αίσθημα δικαιοσύνης, μια αίσθηση δικαίου. Το μέγιστο αίσθημα δικαιοσύνης είναι όλοι να πληρώνουν τους φόρους τους οποίους πρέπει, τους οποίους οφείλει. Και ένα από τα σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο σε επίπεδο δημοσιονομικό αλλά και σε επίπεδο αντίληψης, είναι ότι η φοροδιαφυγή και άλλες μάστιγες αποτρέπουν την ύπαρξη αυτής της αίσθησης δικαίου και ισοτιμίας. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο μέσω των κρατών μελών και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε η διοικητική δομή της χώρας να ισχυροποιηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλοι όσοι πρέπει να φέρουν εις πέρα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις να το κάνουν, έτσι ώστε όλοι να συνεισφέρουν φορολογικά ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Όσο υπάρχει μια μαζική φοροδιαφυγή και απάτη όπως στην Ελλάδα, δεν θα υπάρξει αυτή η αίσθηση δικαίου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές αποφασιστικές και οι επόμενες ώρες είναι τέτοιες. Κεφαλαιόδη σημασία έχουν οι στιγμές αυτές, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για την Ευρωζώνη και ακόμα θα έλεγα ακόμα παρατέρα για τη σταθερότητα της, της παγκόσμιας οικονομίας. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε όλους όσους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην Ελληνική Βουλή να το κάνουν. Να το πράξουν. Όσο μεγαλύτερη ομοφωνία, όσο μεγαλύτερη ενότητα υπάρχει, τόσο το καλύτερο θα είναι για τον ελληνικό λαό και για το μέλλον της Ευρώπης. Σχετικά με το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης, το είπα και το επαναλαμβάνω. Θα ήταν καλό να λήξουν οι εργασίες μας με ένα συμβιβασμό. Προφανώς δεν είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να απευθύνω μια έκκληση μια έκκληση σε αυτή την, στο αίσθημα της, της, του συμβιβασμού θα έλεγα στο οποίο αγκυρώσαμε τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάναμε μέχρι τώρα υπό την Ουγγρική ε, Προεδρία. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε συμφωνήσει στο 98% των διαφορών μας. Έχουμε καλύψει τουλάχιστον το 95% από αυτές. Κάναμε μια τεράστια δουλειά, βελτιώσαμε το κείμενο της Task Force και ταυτόχρονα βελτιώσαμε και τα κείμενα των κρατών μελών. Το τελευταίο κομμάτι ε, μένει να γίνει ακόμα και καλό θα είναι να το ολοκληρώσουμε πριν από τις θερινές διακοπές έτσι ώστε να μπορέσουμε και σε επίπεδο οικονομικής διακυβέρνησης μια ολοκληρωμένη λύση, ένα συνολικό πακέτο, το λεγόμενο Comprehensive Package, το οποίο προτείναμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και λίγους μήνες. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ για το περιεχόμενο της συμβιβαστική λύσης. Αυτό θα το κάνει η Ουγγρική Προεδρία και εσείς φυσικά σαν Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω ότι μετά από τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν, νομίζω ότι θα ήταν κρίμα να μην μπορέσουμε να καταλήξουμε στο τελευταίο 5%. Για το Σέγγεν τώρα. Και εδώ θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία προείπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήμουν παρόν φυσικά στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και όλες οι ευαισθησίες οι οποίες ακούστηκαν εδώ, τις άκουσα και τότε σε αυτό τον γύρο της τράπεζας. Δεν είχα την αίσθηση ότι είχα μπροστά μου 27 δολοφόνους της συνθήκης του Σέγγεν. Δεν ήταν ένα δείπνο δολοφόνων της συνθήκης του Σέγγεν, όχι. Αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε είναι ένα ισόρροπο θα έλεγα πακέτο και η φοβερή αυτή η ρήτρα ασφαλείας αν θέλετε είναι μια ρήτρα την οποία πρότειναν όχι μόνο κάποια αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περιμένουμε και με ε, αγωνία θα έλεγα την τελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε την, ε, τα στοιχεία θα έλεγα αυτής της πρότασης. Όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριελήφθησαν στα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου με συγκεκριμένες αποχρώσεις. Έκανα μια πολύ προσωπική ανάγνωση των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου. Φυσικά το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη μία διασώζουμε το κεκτημένο του Σέγγεν και από την άλλη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες νέες καναστάσεις οι οποίες δεν είχαν απλά προβλεφθεί όταν διαπραγματευθήκαμε τη συνθήκη του Σέγγεν. Από τότε έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει σε βάθος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Και θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για τις νέες προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας και γι' αυτό ε, καταλήξαμε σε αυτά τα οποία γνωρίζετε. Και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συναπόφασης θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχουν καινούριε καταστάσεις δεν μπορούμε παρά να προσαρμόσουμε τις διατάξεις τις οποίες έχουμε ακόμα και όταν είναι τόσο σημαντικές όπως η συνθήκη του Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαν Ρόμπαϊ και για την παρουσίασή σας και για τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Μπαρόσο που μας απίθυνε το λόγο και έδωσε απαντήσεις σε πάρα πολλά θέματα. Κλείνω την συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων ανοιχτή σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.